Καλημέρα σας σε όλες και σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το εξής, μάλλον να σας ανακοινώσω ότι οι σημερινοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν να παρουσιάσουν τις ομιλίες τους με τρόπο ώστε να μείνει ένα δεκάλεπτο μετά από κάθε παρέμβαση για συζήτηση με το κοινό και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και περνούμε αμέσω στα θέματα που έχουμε για σήμερα στη μερίσια διάταξη. Νομίζω ότι μετά από τη χτεσινή πολύ καρποφόρα ημερίδα που ακούσαμε τους πολιτικούς ηθήνοντες, τον εκπρόσωπο της Γαλλομάθειας, εκπροσώπους ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επικεφαλής ε, των υπηρεσιών διερμηνίας διαφόρων διεθνών οργανισμών που μας μίλησαν αφενός για τον λόγο ύπαρξης της πολυγλωσσίας και αφετέρου για την ανάγκη εκπαίδευσης νέων γενεών ε, γλωσσομαθών και κυρίως ε, διερμηνέων συνεδρίων για να εξασφαλιστεί η πολυγλωσσιακή στο μέλλον. Αφού τα κάναμε όλα αυτά χτες λοιπόν, σήμερα θα δώσουμε το λόγο στην έρευνα και στον πανεπιστημιακό κόσμο. Θα μπούμε πρώτα στον συναρπαστικό κόσμο των νέων τεχνολογιών και στη συνέχεια με την άδεια του ε, Πρίτανη στη γνώση της πιο τέλειας μηχανής που υπάρχει, που δεν είναι άλλη από τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον δόκτορα Βάιμπελ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλσρούης αφενός στη Γερμανία, αλλά και στο Πίτσπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών, που χωρίς καμία αφιβολία γνωρίζετε όλοι ότι είναι αυθεντία διεθνώς σε ό,τι αφορά την αυτοματοποιημένη μετάφραση μεταξύ άλλων. Έχετε μέσα στο λόγο, παρακαλώ, κύριε Βάιμπελ. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε Μαρτίνης, κυρία Γενική Διευθύντρια ε, Κοσμίδου, ε, κύριε Διευθυντά, Χωάν Κάρλος Χιμένες Μαρίν, με μεγάλη χαρά ήρθε ενώπιό σας να μιλήσω. Είναι πολύ εντυπωσιακή η ε, ομάδα, το ακροατήριο που έχω την ευκαιρία να μιλήσω, είχα ήδη την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να επισκεφθώ το κοινοβούλιο και να δω τι κάνετε από πλευρά μετάφραση. και επίσης έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους μεταφραστές, συγγνώμη, διερμηνείς, ε, λέει ο, ο διότι ε, διερμηνεύουν σε 24 γλώσσε. Είναι καταπληκτική αυτή η δυνατότητα που έχετε. Εγώ μιλώ πέντε γλώσσες, αλλά δεν θα μπορούσα ότι για τρία λεπτά να κάνω τη δουλειά σας, διότι η συγκέντρωση και η εφράδια που απαιτείται είναι πραγματικά συναρπαστική ανθρώπινη ικανότητα. Τι θα προσπαθήσω εγώ σήμερα να σας παρουσιάσω. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ε, ο στόχος, αφού θα δείτε ότι είναι και αδύνατο άλλωστε, να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο διερμηνέα. Είναι καταπληκτική, απίστευτη αυτή η ικανότητα. Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ να σας πω είναι πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι τεχνολογίες για τους υπολείπους. Εμάς τους υπολείπους θα πρέπει να ε, θυμηθούμε ότι το όνειρό μας για όλους, σε όλο τον κόσμο είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούμε να υποβληθούμε ούτε στην προσπάθεια ούτε στη δαπάνη την οποία ε, υποβάλλεται και μπορεί να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, τούτο εδώ το ακροατήριο γνωρίζει πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό. Εργαζόμαστε ε, όλοι μαζί σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο που και ζούμε. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες, επικοινωνούμε και για την Ευρώπη ανεξάρτητα από τις γλώσσες της, ε, είναι υποχρέωσή της να ολοκληρώνεται. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μιλούμε όλοι την ίδια γλώσσα. Υπάρχει όμως και η αντίθετη ε, τάση ε, ότι προωθούμε και προάγουμε την κάθε γλώσσα, την ομορφιά της, την ταυτότητά της, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Και ο καθένας είναι περήφανος για τη γλώσσα του. Αυτό είναι λοιπόν τώρα μια πρόκληση πώς θα επιτύχουμε αυτό το παγκόσμιο χωριό χωρίς να παραγνωρίσουμε ή να αγνοούμε τις ε, πολιτιστικές μας ταυτότητες. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου που να το καταλαβαίνει αυτό περισσότερο από την Ευρώπη. 24 γλώσσες στην τελευταία καταμέτρηση που έγινε και πολλές διαλέκτους έχει η Ευρώπη και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, αυτή τη στιγμή ε, η κατανόηση είτε δεν γίνεται καθόλου είτε γίνεται με ανθρώπινη διερμηνία. Όλες οι περισσότερες μάλλον διασκέψεις οποίες εγώ πηγαίνω ε, γίνονται σε σπαστά αγγλικά. Κοιτάξτε πώς ομιλούν την αγγλική στην Ευρώπη. Για όσους από εσά πιστεύετε ότι η λύση είναι να το γυρίσουμε στα αγγλικά, κοιτάξτε πώς έχει κατάσταση στις διάφορες χώρες. Μόνο κατά μέσο όρο 30 με 40% των πολιτών ε, ομιλούν αγγλικά αρκετά καλά για να μπορούν να συνεννοούνται σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν το αποκλείουμε ως λύση. Και μάλλον δεν είναι και επιθυμητό έτσι κι αλλιώς. Τι άλλο όμως μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μεταφράσει και διερμηνία, περίπου 500.000 είναι διερμηνεί παγκοσμίω, 150.000 στην Ευρώπη. Διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά η έρευνά μας αυτό το αποτέλεσμα έχει. 31 δισεκατομμύρια δολάρια η αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,3 δις ευρώ ε, δαπανώνται για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνίας. Παγκοσμίως είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία. Στην Ευρώπη έχουμε 24 ε, γλώσσες, είπαμε, στον κόσμο 6.000 και αν ε, ε, μετρήσετε όλους τους συνδυασμούς είναι 36 εκατομμύρια. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε μικρό είναι μόνο το κλάσμα που μπορεί να μεταφραστεί ή που μεταφράζεται. Και είναι κείμενο βεβαίως για ομιλία τα, μάλλον αυτά για τα κείμενα, για τη ε, διερμηνία είναι η κατάσταση ακόμα χειρότερη. 300.000 ε, είναι το χρόνο οι διασκέψεις, το 1% και λιγότερο ε, διερμηνεύεται στο YouTube. Κάθε λεπτό έχουμε 13 ώρες βίντεο που ε, αναρτώνται. Και τηλεόραση, διαλέξεις, ε, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις παράγουν ομιλίες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συναντήσεις, υπάρχει μια σειρά ανθρωπίνων επαφών ε, που γίνονται ανταλλαγές ε, και δεν μπορεί ο ένας να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του άλλου. Τι μπορεί να γίνει τώρα. Είναι τεράστια η πρόκληση και δεν μπορεί πιστεύω να αντιμετωπιστεί μόνο και αποκλειστικά από την ανθρώπινη προσπάθεια. Γι' αυτό αφιερώνουμε πολύ χρόνο, προσπάθεια και χρήμα για να βρούμε αυτόματες λύσεις. Μπορεί όμως η τεχνολογία να δώσει λύση. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η προσπάθεια, η μετάφραση, η διερμηνία ε, μιας ομιλίας από τη μία γλώσσα στην άλλη. Επί μία εικοσαετία και πλέον εργαζόμαστε στο πρόγραμμα και το πρόβλημα αυτό και ουσιαστικά και χοντρικά έχουμε τρία διαφορετικά βήματα σε δύο κατευθύνσεις. Αν θέλουμε να μεταφράσουμε από τα αγγλικά στα ισπανικά, το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι σύστημα να αναγνωρίζει την ομιλία και να ε, κάνει ε, τον προφορικό λόγο γραπτό. Το δεύτερο θα είναι ένα σύστημα μετάφρασης που θα μεταφράζει το κείμενο, το κείμενο από τα αγγλικά στα ισπανικά και από την άλλη χρειάζομαι και ένα σύστημα το οποίο να ε, εκφέρει προφορικά την ισπανική ομιλία για να το ακούσει ο ισπανόφωνος και όταν θέλει να απαντήσει χρειαζόμαστε την αντίστροφη διαδικασία αναγνώριση της ισπανικής ομιλίας μετάφραση του γραπτού κειμένου και εκφορά του προφορικού στα αγγλικά αυτό έχει λειτουργήσει για πολλά χρόνια και μόλις πρόσφατα την τελευταία δεκαετία καταλάβαμε ότι είναι αδύνατο να προγραμματίσει κάνει ένα τέτοιο σύστημα γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί κανόνες για να κατανοηθεί η ανθρώπινη γλώσσα. Γι' αυτό όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βασίζονται σε τεχνικές αυτόματης εκμάθησης. Οι μηχανές μας που θα σας παρουσιάσω εκπαιδεύονται με βάση δεδομένα με τρόπο αυτόματο. Το διαδίκτυο ε, δίνει στοιχεία σε πολύ μεγάλο όγκο, όλο και περισσότερο και μπορούμε να απευθυνθούμε εκεί, να συλλέξουμε στοιχεία παγκοσμίω ε, έτσι ώστε να έχουμε βάσεις δεδομένων για να εκπαιδεύσουμε αυτόματα τα συστήματα. Ε, συλλέγουμε λοιπόν δεδομένα από ομιλίες και από μεταφράσεις και έτσι οι μηχανές μας μαθαίνουν και βελτιώνονται συνεχώς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούν αυτά τα μοντέλα, απλώς σκεφτείτε ότι είναι λεξικά ε, και συλλογική μνήμη, ας πούμε, που συλλέγει ε, στατιστικές και μαθαίνει πώς μεταφράζεται μια λέξη και πώς χρησιμοποιείται σε ένα γλωσσικό πλαίσιο σε κάθε μία από τις καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει. Με αυτές τις τεχνικές, λοιπόν, διανύσαμε ε, τέσσερις φάσεις στην έρευνα μας. Ε, τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχή της δεκαετίας του 90 ε, άρχισαν τα πρώτα συστήματα που ήταν λειτουργικά. Ο Ιανός ήταν το πρώτο σύστημα στην Ευρώπη, όπου είχαμε 200 έτοιμες προτάσεις και χρειαζόταν πέντε λεπτά για να βγει από την άλλη πλευρά μία φράση από τις 200. Αλλά έπρεπε να είμαστε βέβαιοι ότι ήταν σωστή και η σύνταξη και ε, το λεξιλόγιο ήταν 100 με 200 λέξεις. Ε, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ πρακτικό. Την επόμενη δεκαετία ε, δημιουργήσαμε αυθόρμητα συστήματα. Όταν κάποιος μιλάει μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε το ύφος, ούτε ο τόνος, ούτε το λεξιλόγιο. Διστάζουμε όταν μιλούμε. Όλα αυτά θα πρέπει να τα χειριστεί και η μηχανή και να τα καταλάβει. Ευτυχώς από όλα αυτά βγήκαν δύο κατευθύνσεις που μπορούμε σήμερα να εφαρμόσουμε στον πραγματικό κόσμο. Το ένα ε, είναι κινητές ε, συσκευές ας πούμε επακολουθητικής διερμηνίας. Είναι σημαντικό αυτό για ταξιδιώτες, για ανθρωπιστικές αποστολές, για επαγγελματίες της υγείας, ε, για στρατιωτικούς, ε, αστυνομικούς, ε, κυβερνητικές επιχειρήσεις όπου κάποιος πρέπει να δράσει επιτόπου με κινητές μονάδες. Και το δεύτερο είναι ε, ταυτόχρονη διερμηνία ε, σε μη μετακινούμενο περιβάλλον, ας πούμε ειδήσει, ε, τηλεόραση, κυβερνητικές ομιλίες, πανεπιστήμια. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τις δύο πρώτες συσκευές. Τι θέλουμε, είμαστε κάπου επιτόπου και θέλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας και το σύστημα αυτό να το μεταφράσει ή να το διερμηνεύσει στην άλλη γλώσσα και να μπορέσει και ο συνομιλητής σας να απαντήσει στη δική του γλώσσα και να απευθυνθεί σε εσά. Αυτό το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό για ανθρωπιστικές αποστολές όπου στο παρελθόν χρησιμοποιούσαμε ανθρώπους για τη διερμηνία αλλά πολύ συχνά σε περιοχές κρίσεων ε, δεν έχουμε διερμηνείς. Γι' αυτό Προσπαθούμε με ε, κάποια διαγράμματα, με κάποια λεξικά να εργαστούμε, αλλά είναι προβληματικό, διότι δεν ε, μπορεί να γίνει διερμηνία με τέτοιο τρόπο. Και επίσης υπάρχουν και θέματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε και ποιο μεταφραστή ή διερμηνέα θα βρούμε και αν είναι αξιόπιστη η μετάφραση και η διερμηνία τόπου. Τι κάναμε λοιπόν. Και πάλι έχουμε αναπτύξει συστήματα ε, για ταξιδιωτικούς σκοπούς και δημιουργήσαμε και συστήσαμε μια μικρή εταιρεία που προσπαθεί αυτό να το ε, μεταφέρει σε μια προσιτή τιμή να μπορούμε όλοι να αγοράζουμε αυτές τις συσκευές ε, και να το κατεβάζουμε στο τηλέφωνο μας ως εφαρμογή από ένα App Store. Η εταιρεία μας λοιπόν και ε, το λογισμικό λέγεται GBCO και μπορείτε να το κατεβάσετε στο Android ή στο iPhone. Ε, έχει 10 γλώσσες, με 15 αυτή τη στιγμή, 40.000 ε, λέξεις, λύματα και επίσης δεν χρειάζεται διαδίκτυο, ε, αρκεί το τηλέφωνο. Αυτό είναι σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό ε, για ανθρωπιστικές αποστολές, γιατρούς, στρατιωτικούς κτλ. Γιατί ε, δεν έχουμε σε τέτοιες καταστάσεις επιτόπου διαδίκτυο πάντα. Αυτό είναι λοιπόν εδώ το σύστημα. Είναι μια εφαρμογή, ένα app που κατεβάζετε στο iPad, στο iPhone και μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα το διώνυμο της γλώσσας και άρεσε τόσο πολύ αυτό στην Apple που προς μεγάλη μας χαρά έκαναν διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Ιαπωνία. After college and with my iPhone, I checked out hostels before booking them. Shared pictures as I went. My mom loved that. And I even downloaded this app which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. So we were, of course... Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ με τη διαφήμιση αυτή, αλλά όπως βλέπετε, για να δείτε μάλλον ότι λειτουργεί, σας έφερα και το δικό μου iPad και μπορείτε να διαβάσετε καλύτερα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 So, with these devices we have... Βλέπετε ότι με αυτές τις συσκευές έχουμε επεκταθεί σε διάφορες άλλες συσκευές και βλέπετε ότι κάνουν και λάθη. Και ε, αφιερώνουμε πάρα πολύ προσπάθεια για να διορθώνουμε τα λάθη αυτά. Και βέβαια και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και ακριβώς μία από τις συναρπαστικές πραγματικά ιδιότητες που έχουμε είναι να διορθώνουμε τα λάθη μας. Ενώ αυτές οι συσκευές ή καν κακή μετάφραση ή σφάλμα μπορούμε να, το, να τις ε, ε, ε να τις αλλάξουμε, να γράψουμε το κείμενο ε, για να διορθώσουμε. Μαθαίνουμε και από τις διορθώσεις αυτές, γιατί κάθε φορά που κάνουμε μια διόρθωση έχουμε νέα στοιχεία και βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας. Αυτά τα συστήματα τα εφαρμόζουμε και σε ανθρωπιστικές ε, αποστολές κάθε χρόνο σε τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου. Βλέπετε εδώ καταστάσεις όπου χρειαζόμαστε τέτοια μηχανήματα, όπου υπάρχουν μεν διερμηνείς, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Εδώ βλέπετε έναν από τους γιατρούς ε, που στην Ταϊλάνδη χρησιμοποιεί το μηχάνημα αυτό σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της νότιο-ανατολικής ε, Ασίας και με ιατρικά πολιτικά προγράμματα ε, κάνουν δοκιμές για το πώς μπορεί να γίνει ε, μια καλύτερη πολιτική προστασία και προσπαθούμε λοιπόν κάθε χρόνο στην Ταϊλάνδη σας δείχνω την άσκηση στην Ταϊλάνδη και στην Καμπότζη και πάντα εκεί έχουμε ε, γλωσσικά προβλήματα. Κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμος ε, δέχεται ιατρική βοήθεια και επειδή καραδοκούν γλωσσικά προβλήματα χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές. Να, εδώ μια άλλη φωτογραφία από μια ανθρωπιστική ε, αποστολή του Πίτσμπουργκ στη Νότια Αμερική, στη Ονδούρα. Μια κλινική από το Pittsburgh έχει ένα πρόγραμμα ε, με γιατρούς όμως που δεν μιλούν ισπανικά και παίρνουν τις συσκευέ μας επιτόπου για να μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με τους ασθενείς τους σε αυτό το πρόγραμμα shoulder to shoulder. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται πολύ μεγάλη ε, προσπάθεια και βελτιωνόμαστε και ελπίζω να σας έπεισα ότι σε όλες αυτές τις καταστάσεις δεν μπορούμε πάντα να περιμένουμε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα διερμηνέα άνθρωπο. Ακόμα και αν ε, υπολείπονται φυσικά οι μηχανές, ε, είναι πολύ σημαντικό να τις έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούμε αυτό σε ανεπίσημα κανάλια, όχι πάντα σε επίσημους διάβολους ε, την ε, κυβερνητική συνδρομή. Όπως βλέπετε τώρα έχουμε και ε, ταυτόχρονη μετάφραση, η διερμηνία. Όταν βλέπει κανείς τηλεόραση, έχουμε διαλέξεις, κοινοβουλευτικές μιλίες, τηλεφωνικές διαλέξεις, πανεπιστημιακούς είναι συνεχής η ροή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να πατήσει κάποιος ένα κουμπί, να σταματήσει τη φράση, να την επαναλάβει κτλ. Είναι μια ομιλία που ρέει. Βεβαίω έχουμε πολλά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε πάνω σε αυτά να βασιστούμε και να επεκτείνουμε και να βελτιώνουμε τα συστήματά μα για ταυτόχρονη ε, διερμηνία. Ε, τώρα, σε πανεπιστημιακές διαλέξεις έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι Εκεί δεν έχουμε διερμηνείς ανθρώπους, αλλά φοιτητές που δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, γερμανικά στο πανεπιστήμιό μας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να τους δίνουμε τα εργαλεία για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν μία διάλεξη στα γερμανικά και να καταλάβουν το περιεχόμενό της. Άρα έχουμε κάποιον που νομίλει μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε και βεβαίω είναι πρόκληση αυτό και θέλουμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα στον ακροατή να καταλάβει το περιεχόμενο. Τα αυτόματα συστήματα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να είναι όσο καλή μπορεί να είναι σήμερα η ανθρώπινη μετάφραση ή διερμηνία. Αλλά φανταστείτε, είστε σε μια χώρα που δεν παρέχονται υπηρεσίε διερμηνία και δεν καταλαβαίνετε γρή. Λοιπόν, δεν θα προτιμούσατε να έχετε ένα σύστημα που να σας βοηθάει λίγο, να σας δίνει λίγη δερμηνία να μπορέσετε τουλάχιστον να παρακολουθήσετε την ουσία, την κεντρική ιδέα της διάλεξης. Μας λέγουν λοιπόν οι φοιτητέ μας ε, στη Γερμανία ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς, ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο να μάθουν γερμανικά παρά να μάθουν το αντικείμενο που ήρθαν να σπουδάσουν. Και ε, κάνουν μαθήματα γλώσσας πριν ε, έρθουν στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως δεν θέλουμε εμεί να του αποθαρρύνουμε να μην μάθουν γερμανικά. Θέλουμε να του ενθαρρύνουμε να μάθουν γερμανικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ε, διαφυγή εγκεφάλων. Και θέλουμε ε, να έρχονται στη Γερμανία ακόμα και αν υπάρχει αυτός ο γλωσσικός φραγμός. Χρηματοδότηση. Παίρνουμε βεβαίως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ένα πρόγραμμα που λέγεται U-Bridge, όπου υπηρεσίε μετάφραση και διερμηνία αναπτύσσονται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και παρέχονται και υπηρεσίες γενικότερα. Το σύστημα τα συστήματα που βλέπετε εδώ έχουν αναγνώριση και μετάφραση, αλλά εκτός αυτού έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα ότι όταν εκφέρω ε, ε, εγώ μια πρόταση δεν λέω τελεία ή κόμμα και πρέπει η μηχανή να καταλάβει πού τελειώνει η πρόταση για να κάνει τη μετάφραση. Ε, αυτός ο συνεχόμενος μονόλογος λοιπόν είναι μια επιπλέον πρόκληση για τη μηχανή μετάφραση. Το δεύτερο πρόβλημα είναι και πώς φτάνει το αποτέλεσμα ακουστικά στα διάφορα μέλη του ακροατήριου. Όλοι μιλούμε γλώσσες και τις ακούμε, αλλά μπορούμε κάποια στιγμή ο καθένας να έχει την προσωπική του συσκευή μετάφρασης ε, και να ε, φτάνει ατομικά στον κάθε ακρότη η μετάφραση με διαφορετικό τρόπο. Τι κάνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο της Καλσρόης. Ένα σύστημα το οποίο μεταφράζει μέσω του διαδικτύου και ο τρόπος ε, να φτάνει το μήνυμα σε όλους είναι το διαδίκτυο. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, κάνει μια διάλεξη, ομιλία, πηγαίνει σε ένα σερβερ, σε έναν υπολογιστή, στον υπολογιστή αναγνωρίζεται, μεταφράζεται στην άλλη γλώσσα και μετά ε, με μια ιστοσελίδα φτάνει στον φοιτητή. Φέρνει ο φοιτητή το λάπτοπ του ή δεν ξέρω τι συσκευή του και παρακολουθεί το περιεχόμενο και τη μετάφραση, το γραπτό, προσωπικά ο καθένας. Μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία ε, θα μεταφράζεται και το παρακολουθεί στην οθόνη του. Αυτό γίνεται με ε, σερβες που έχουμε στο πανεπιστήμιο και μπορεί να μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Το καλοκαίρι το κάναμε ε, σε τέσσερα μαθήματα από τα γερμανικά στα αγγλικά. Κάνουμε και άλλα όμως. Ε, μεταφράζουμε αυτόματα τις διαφάνειες PowerPoint που δείχνουμε στο μάθημα έτσι ώστε οι φοιτητές που δεν καταλαβαίνουν στα γερμανικά τη διαφάνεια να την έχουν μεταφρασμένη στα αγγλικά. Μετά ε, τη διάλεξη μπορούν να τη βρουν στο σερβερ και να ξανακούσουν ή να διαβάσουν ε, τη διάλεξη μετά το τέλος της ε, βάσει του αρχείου που έχουμε και ε, μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα αναζήτησης, επανάγνωσης. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μια λέξη κλειδί και με βάση αυτή τη λέξη να βρει τη διάλεξη και να την ξαναδιαβάσει. Ποιε είναι τώρα ακόμα οι προκλήσει που έχουμε για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα. Όπω ε, όπως σας είπα προηγουμένω, είναι ένα συνεχιζόμενος μονόλογο. Δεν λέμε τελεία ή κόμμα. Επίση το ύφο είναι αυθόρμητο, κατακαιρματισμένο, γρήγορο πολλέ φορέ. Ε, καμιά φορά Κανεί μπορεί να βύχει, να γελάει κατά τη διάρκεια του μαθήματο, ακόμα και να τραγουδάει. Όλα αυτά χρειάζονται επεξεργασία. Επίση, το λεξιλόγιο μα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια σε επίπεδο διάλεξη στο Πανεπιστήμιο είναι πολύ ορολογία. Γι' αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις διάφορες λέξεις που εμφανίζονται σε διάφορες διαλέξεις και μου ζήτησαν οι διερμηνείς εδώ στην αίθουσα να τους δώσω τις διαφάνειες για να προετοιμαστούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να προσαρμόζουμε πάντα το λεξιλόγιο, να ευθυγραμμίζουμε το ανθρώπινο στο λεξιλόγιο της μηχανής. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Και υπάρχει και πρόβλημα πάλι και για τον άνθρωπο διερμηνέα αλλά και για τη μηχανή να το κάνει με πολύ μεγάλη χρονική υστέρηση για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί ταυτόχρονα τη διάλεξη. Τα γερμανικά για μας ήταν ιδιαίτερη πρόκληση. Όσοι από σας γνωρίζετε γερμανικά ξέρετε ότι ε, έχει αυτό το πρόβλημα, το δυσάρεστο, η γλώσσα που το ρήμα έρχεται στο τέλος και πρέπει να περιμένεις ένα λεπτό για να δεις πώς θα τελειώσει η ιστορία και έχουμε και τις καταλήξεις και όλα αυτά τα σύνθετα ε, ε, ουσιαστικά που πρέπει να ε, τα κόβουμε. Ε, ας πούμε, μια, λέξη μια έννοια που είναι τέσσερις λέξεις στα αγγλικά, στα γερμανικά είναι μία. λοιπόν, είπαμε, η ορολογία για ένα τεχνικό θέμα. Επίσης, έχουμε και μαθηματικούς τύπους. Όταν κάποιο μιλάει για ένα μαθηματικό τύπο, δεν μπορεί να το μεταφράσει, πρέπει να το δει γραμμένο. Και υπάρχει ε, και το θέμα της αμφισημία. Το προσ... Η λέξη Vorzeichen στα γερμανικά μπορεί να σημαίνει πρόσημο, θετικό ή αρνητικό ή μπορεί να σημαίνει και ε, ιονός. δεν ξέρει κανείς κάθε φορά τι είναι αυτό. Επίσης, πολλές φορές ε, ε, παρισφρίουν αγγλικές λέξεις σε άλλες γλώσσες. iPhone, iPad, laser και ε, στα γερμανικά σε μια διάλεξη προφέρονται με την αγγλική τους προφορά. Ή όταν λέμε download, στα γερμανικά κλείνεται η λέξη αυτή όπως ένα οποιοδήποτε γερμανικό ρήμα. Λέμε downloaded, δεν λέμε downloaded. Ε, είναι τεράστια λοιπόν αυτή η πρόκληση για το μηχάνημα, για να καταλάβει τι κάνουμε, αλλά και για τον άνθρωπο. Ε, χρειάζεται συνεχής προσαρμογή. Για τα μηχανήματα έχουμε συνεχή προσαρμογή και αναπροσαρμογή των συστημάτων και χρησιμοποιούμε και τις διαφάνειες του PowerPoint και οι υπολογιστές μας για να βρουν όλη αυτή την ορολογία που χρησιμοποιούμε μέσα στις διαφάνειες με ε, μια ορολογία που ψάχνουμε και στο διαδίκτυο για αντίστοιχα κείμενα και από τα κείμενα αυτά αναπαράγουμε όλες αυτές τις λέξεις για να τις βάλουμε στο σύστημα. Τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι Πώς θα φύγουμε από αυτή την κατάσταση για να τη μεταφέρουμε σε 6.000 γλώσσε στον κόσμο. Κάνουμε πάρα πολλή έρευνα για να ε, φθηνίνει αυτή η διαδικασία και να γίνει πιο αποτελεσματική με νέα συστήματα, ακόμα και για άλλες γλώσσες που δεν έχουν τόσα χρήματα. Μου κάνουν νόημα ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Συμπέρασμα. Είναι δυνατή διερμηνία ε, με μηχανήματα. Ναι, πιστεύουμε εμείς και θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται μαθαίνουν από στοιχεία ε, και δεδομένα του διαδικτύου. Όσο περισσότερα στοιχεία έχει το διαδίκτυο, τόσο θα βελτιώνονται τα μηχανήματα και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δεδομένα. Θα αντικαταστήσουμε ε, τους ε, ανθρώπους διερμηνείς. Όχι, και το λέω αυτό με πάθος. Η ποιότητα της μηχανικής μετάφρασης παραμένει πάρα πολύ χειρότερη και επίσης να έχει την ανθρώπινη κρίση και διέστηση για να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Ε, ωστόσο, δεν είναι αυτό τώρα ανταγωνισμός ανθρώπου-μηχανήματος. Οι υπόλοιποι, εμείς τι κάνουμε, που δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε την ευκαιρία να χαιρόμαστε πάντα να απολαμβάνουμε τις θαυμάσιες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνίες σας. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ποια είναι η πραγματικότητα κακά αγγλικά ή καθόλου επικοινωνία. Ε, και αυτό είναι πραγματικά κοινωνική πρόκληση. Τι θέλουμε να γυρίσουμε στο μεσαίωνα που μόνο οι μορφωμένοι καταλάβαιναν τι έλεγε η κυβέρνηση και η εκκλησία. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε μετάφραση για όλους και για τους αυτούς μας. Ε, εμποδίζουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ακούει ο κόσμος τι έχει να πει ο άλλος και σιγά σιγά ενδιαφέρεται και παροτρύνεται να μάθει και μια άλλη γλώσσα. Και το έχουμε δει και αυτό. Ορισμένα από τα μηχανήματά μας χρησιμοποιούνται από το κοινό ακριβώς για να μάθουν την άλλη γλώσσα. Ποια είναι λοιπόν η αποστολή μας. Να έχουμε ε, πολύγλωση, ε, κατανόηση και ε, ένταξη και ολοκλήρωση όλων, να διατηρήσουμε τη γλωσσική μας πολυμορφία κληρονομιά και να την ε, τροφοδοτούμε. Ε, και θα πρέπει η Ευρώπη να το αναλάβει αυτό και όχι να το αναθέσει σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλες εταιρείες. Μόνοι μας να το κάνουμε. Επίσης, για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ε, αγκαλιάσουμε και να εστερνιστούμε και την ανθρώπινη και τη μηχανική υποστήριξη. Και τα δύο πιστεύουμε ότι χρειάζεται γι' αυτό συμβίωση με ε, λύσεις ε, που να ε, συμπληρώνουν και να μεγεθύνουν την ανθρώπινη προσπάθεια με μηχανική υποστήριξη. Ελπίζω να σας έδωσα μία γεύση για το τι αναμένετε και πραγματικά σε αυτή τη συμβίωση ποντάρουμε και από εκεί θα έρθει η λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, δόκτωρα Βάιμπελ. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Αντιπρόεδρος ε, ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του, αλλά ε, δεν μπόρεσε να μείνει άλλο στην διάσκεψη, έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει. Ήρθε η ώρα για τη συζήτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες, σχόλια. δεν ξέρω αν η μηχανή σας το μάκι ε, θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Πάντως, αν κάποιος θέλει το λόγο, ας το κάνει τώρα ή ας το πάσει για πάντα. Η Εμπρού. Σας ευχαριστώ. Ήταν καταπληκτική η ομιλία σας. Έχω μια ερώτηση για την πρόληψη. Γιατί μιλήσατε για δύσκολες γλώσσες όπως τα γερμανικά, τα τουρκικά είναι ακόμη χειρότερα. Γιατί θα πρέπει να αναλύσει κανείς μία λέξη που είναι πολύ σύνθετη. Είπατε ε, μία λέξη στα γερμανικά αντιστοιχεί στη μετάφραση σε ε, στα γερμανικά αντιστοιχεί σε τέσσερις στα αγγλικά. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Αυτό είναι το πρόβλημα των σύνθετων λέξεων στα γερμανικά. Ξέρετε την ε, περίφημη ιστορία. Ο, ο καπετάνιος της εταιρεία που έχει πλοία πάνω στο Δούναβι, όλα αυτά είναι μία λέξη στα γερμανικά και είναι ανέκδοτο στα γερμανικά. Ε, και έχουμε και πτώσεις και κλήσεις και για να το μεταφράσουμε θα πρέπει να σπάσουμε στα σύνθετα της αυτή τη γλώσσα. Και ε, στα τουρκικά είναι αυτή η μορφολογία αντίστοιχη και τεράστιο πρόβλημα. Ε, αναλύουμε τα μορφώματα και στα ε, Ιαπωνικά και στα Ρωσικά είναι αυτό ε, και θα πρέπει να σπάσουμε όλες τις προτάσεις για να τις μεταφράσουμε και μετά να τις συνενώσουμε για να βγει το τελικό αποτέλεσμα στην άλλη γλώσσα. Άρα πρώτα έρχεται το κείμενο. Δηλαδή η ομιλία γίνεται κείμενο, αναλύεται και μετά συντίθεται. Δεν είναι όπως ε, η ανθρώπινη διερμηνία που εκ των προτέρων υποθέτουμε κάποια πράγματα. Ναι. Ναι, προσπαθούμε να τα συνθέσουμε. Δηλαδή το να ε, μαντέψεις ποιο είναι το ρήμα είναι τεράστιο πρόβλημα. Ας πούμε, ε, θέλω να γραφτώ για μία ε, ομιλία που θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα. Αλλά το θέμα αν θα γραφτεί ή αν θα ακυρώσει την εγγραφή σου, το καταλαβαίνει μετά από πέντε λεπτά όταν θα έρθει ε, ε, το πρόθεμα. Γιατί είναι αν μέλντεν γράφομαι, up μέλντεν ε, ακυρώνω την εγγραφή μου. Ξέρουν ε, ξεγράφομαι, α πούμε, ναι. ε, τα ξέρουν αυτά οι διερμηνείς. Αν μαντέψεις λάθος, τελικά, ε, θα πρέπει να το αναθεωρήσεις, να πεις ναι, δηλαδή εννοώ, ξέρετε, και τα λοιπά. και αυτό είναι μια δυνατότητα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνουν το περιεχόμενο και στη συνέχεια έρχονται να διορθώσουν το λάθος τους. το μηχάνημα δεν μπορεί να το κάνει. Και τι συμβαίνει, χάνεται ε, το πρόθεμα στο τέλος εντελώς, δεν αναφέρεται και μένει ελλειπής η πρόταση. Και είναι λάθος αυτό. Και για ένα διερμηνέα επίση είναι και θέμα μνήμη και πρόβλημα. Πρέπει κανεί να θυμάται 10 λεπτά ομιλίας πριν το αναπαράγει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα όμω για τη μηχανή. Γιατί εκεί μπορούμε να ε, αποθηκεύσουμε ώρες ολόκληρε αν θέλετε ομιλιών. Και πάλι επανερχόμαστε στη συμβίωση και στην αλληλοσυμπλήρωση. Υπάρχουν μερικά πράγματα που κάνουν πολύ καλά οι μηχανέ και κάποια άλλα που κάνουν πολύ καλά οι άνθρωποι. Έτσι χρειάζεται λοιπόν συμβίωση και συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις από την Αγία, από την Αγία πολύ Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία και η παρουσίαση. Και καταλαβαίνουμε ότι η διερμηνία μέσω συσκευή είναι κάτι αναπόφευκτο. Μπορεί να είμαστε κατά, μπορεί να μας στεναχωρεί αυτό το γεγονός, είναι μάλλον αναπόδραστη και αυτή η τεχνική εξέλιξη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κάποια ειδικά τεχνικά προβλήματα που μας αναλύσατε και κάποια γλωσσικά. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει μέσα σε 5-10 χρόνια, 10 χρόνια το αργότερο. Τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε μέσα σε 10 χρόνια στην προσπάθεια μετάφρασης, αυτόματης μετάφρασης και αυτόματης διερμηνίας. Είπατε ότι θα αυξηθεί η επιθυμία για εκμάθηση γλωσσών χάρη στην εκτεταμένη χρήση της αυτόματης διερμηνίας. Δεν συμφωνώ όμω ε, μαζί σας. Πιστεύω ότι η μηχανική αυτή μετάφραση ή διερμηνία θα δημιουργήσει μια ψευδέστηση εύκολης επικοινωνίας, αποθαρρύνοντας για την πραγματική εκμάθηση γλωσσών. Η πραγματικότητα είναι περίπλοκη. Όπως και με τις ε, νευρολογικές διαδικασίες βλέπουμε τι αλλαγές ε, ε, παρουσιάζονται στον εγκέφαλο με την εκμάθηση των γλωσσών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα προσπαθήσουμε να τα συμφιλιώσουμε όλα αυτά και να τα συμβιβάσουμε. Δηλαδή, ναι, με να μην εμποδίσουμε ή να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να, μάθουν, να μάθει καλά τη μητρική του γλώσσα και ξένες γλώσσες και ταυτόχρονα να βρούμε μια ισορροπία και μια σωστή λειτουργία για την αυτόματη μετάφραση και διερμηνία. Γιατί και η, ε, η μετάφραση και η διερμηνία από άνθρωπο θα τροποποιηθεί στο μέτρο που εξελίσσεται και η μηχανική και αυτόματη μετάφραση και διερμηνία. Δεν θα είναι ίδια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με αυτά που θα έχουμε μετά από 10 χρόνια. Όταν ετοιμάζουμε λοιπόν τις νέες γενιές διερμηνέων, θα πρέπει να δούμε πώς θα τους προετοιμάσουμε για να εργάζονται στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευκαιρία για τέτοια διερμηνία εκεί που είναι εύχριστο, πρακτικό και φθηνό. Γιατί ε, και η διερμηνία είναι απαραίτητη, γιατί ο άνθρωπος διερμηνέας ε, γνωρίζει καλύτερα το περιεχόμενο, κατανοεί καλύτερα, ενώ οι μηχανές, οι συσκευές αυτές, ε, όπως είδατε, μεταφράζουν με μηχανικό αυτόματο τρόπο και φυσικά κάνουν λάθη. Σε καμία περίπτωση μια συσκευή δεν θα είναι τόσο καλή όσο ένας άνθρωπος, ούτε θα είναι τόσο εκλεπτισμένη η εκφορά ε, του λόγου από έναν άνθρωπο διερμηνέα. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν καλύτερα το περιεχόμενο, τι συγκεκριμένε ομιλίε από ότι μηχανές. Αλλά στα, στη διπλωματία και κάποια, σε κάποιες ε, ειδικέ ε, αποστολές, ανθρωπιστικές αποστολές, φυσικά ο κόσμος προτιμά τον άνθρωπο διερμηνέα. Γιατί ο άνθρωπο διερμηνέα δεν είναι μόνο μηχανή διερμηνία, είναι και βοηθό. Εξασφαλίζει την επικοινωνία, τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Σίγουρα οι ικανότητε του ανθρώπου είναι πολύ ευρύτερε από ό,τι τη μηχανή. Και σε ό,τι αφορά την μελλοντική κατάρτιση, εγώ θα έδινα έμφαση και για τη διερμηνία, στην ποιότητα, στο πλαίσιο της αποστολής του διερμηνέα και του συνόλου του έργου του. Τώρα, αλλά για ανάγνωση εφημερίδας ή παρακολούθηση τηλεόρασης, ε, δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε ένα διερμηνέα δίπλα μας ή στις διαλέξεις των πανεπιστημίων. Δεν μπορούμε να έχουμε 10 διερμηνεί για κάθε διάλεξη. Αν πρότεινα κάτι τέτοιο θα προκαλούσε το γέλο τα, στα γραφεία και στις διοικητικές μας υπηρεσίες. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αλλά οι μηχανές βοηθάν. Τουλάχιστον να έχουμε μια ιδέα του τι διαμείβεται κάθε φορά. Τώρα, δεν πιστεύω ότι με την αυτόματη μετάφραση θα αποθαρρυνθεί ο κόσμος από την εκμάθηση των ξένων γλώσσων, γιατί μαθαίνει κανείς μια γλώσσα όταν τον ενδιαφέρει ένας πολιτισμός και συνήθω ε, πηγαίνει για να γνωρίσει ένα πολιτισμό και όταν θέλει να ταξιδέψει κάπου αισθάνεται πολύ μεγαλύτερο φόβο όταν δεν γνωρίζει τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Όταν κάποιο μπορεί να ταξιδέψει έχοντα μια συσκευή, οπότε κάνει το πρώτο βήμα και αρχίζει και κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον, ενισχύεται και το ενδιαφέρον του να έρθει πιο κοντά στον συγκεκριμένο πολιτισμό και να μάθει και τη συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό ευελπιστούμε ως εξέλιξη. Η Ελίζαμπετ Κρόλ από την Άρτα. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά ομιλούμενη γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από την γραπτή. Υπάρχει η φράση και η μελωδία της φράσης. Εγώ πολύ συχνά δουλεύω από τα γερμανικά και πολύ συχνά μπορούμε να προβλέψουμε χάρη στην ε, μουσική της φράσης ή να φανταστούμε αν υπάρχει άρνηση στο τέλος. Ε, επιτρέπει αυτό να προβλέψουμε και είναι μια διάσταση την οποία δεν μπορεί να λάβει υπόψη η συσκευή. Η μετάφραση γίνεται εδώ σαν να ήταν ένα γραπτό κείμενο ε, που έχει και είναι και επεξεργασμένο και ίσως σε αυτή την άλλη διάσταση να έγκυται μια ενδεχόμενη λύση. Ναι, ναι πολύ σωστή παρατήρηση. Θα ήθελα να σας πω για άλλο ένα πρόβλημα που είναι ακόμα πιο αφηρημένο γιατί είναι η δισταγμή οι μηχανέ, τα συσκευέ, έχουν τεράστιε δυσκολίε να το καταγράψουν αυτό. Αν ήθελα να καταγράψω τις τηλεφωνικές σα συνδιαλέξει με την οικογένειά σα και προσπαθούσα να τις μεταγράψω, και αν έπρεπε να διαβάσουμε αυτό το, την ε, μεταγραφή χωρίς κανένα λάθος και χωρίς καμία παύση, θα σκεφτώσουν ότι ο κόσμος που το έκανε αυτό είναι, θα ήταν μεθυσμένος, γιατί θα δείτε ότι ένα σωρό δισταγμοί υπάρχουν, επαναλήψεις, ε, ερωτηματικά δισταγμοί, ενώ σε ένα αναγνώσιμο κείμενο αυτά εξαφανίζονται. Συν αυτό που είπατε, ότι η, προφορά, η μελωδία της πρότασης ε, που γεννούν επιπλέον προκλήσεις. Αυτά κάπως τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να βρούμε ε, σημεία όπου θα πρέπει να πάει η τελεία και για να μπορέσουμε να βρούμε μια κεντρική δομή. Αλλά είναι ένα ακόμα επίπεδο περιπλοκότητας ε, στο το οποίο ερευνούμε. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις τις αποχρώσεις και την αίσθηση μιας ε, πρότασης, πώς ε, αντιλαμβάνεσαι, πώς πιάνεις το ε, δραματικό, την κίνηση, την μελωδία. δεν, έχουμε, δεν το έχουμε καταφέρει. Πάντως ξέρουμε τις ιδέες, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα όσα περιλαμβάνει η ανθρώπινη ομιλία. Θα πρότεινα τώρα να δώσουμε σε δύο ακόμη ομιλητές στο λόγο και μετά να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Σάλι Μπέιλι από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Κατάλαβα ότι αυτό ισχύει μόνο σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις, περιστάσεις, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο παρουσιάσατε, όπου εγώ διερωτώμαι αν η χρήση των μηχανημάτων αυτών είναι βλαβερός και πρόκειται για την περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, όπου προσπαθούμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί σωματικά να μιλήσουν σε γιατρούς. Πώς μπορεί ένα παιδί να μιλήσει σε έναν γιατρό μέσω ενός μηχανήματος. Μήπως τελικά εμποδίζει την επικοινωνία. Δηλαδή η διερμηνείς είναι τόσο σημαντική για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας που εγώ θα ανέμενα σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλετε καν να χρησιμοποιήσετε μηχανήματα. Ε, είμαι ευτυχής που θίξατε αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε και εμεί την ίδια ανησυχία και φόβο. Δύο πράγματα έχουν γίνει. Καταρχήν αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε μονόγλωσσους τοπικούς ανθρώπους που λειτουργήσαν, που ενεργούσαν ως διευκολυντέ, ε, μεσολαβητές και βοηθοί. Έχετε δίκιο ότι ένας Αμερικανός ε, πεζονάύτη, όταν στέκεται μπροστά σε μια καημένη κυρία στην Ταϊλάνδη είναι τρομακτικό θέαμα. Απ' την άλλη έχουμε Ταϊλανδούς ή Καμποτζιανούς που εργάζονται με τους, λαούς, με τους, με τους ε, ανθρώπους, αλλά είναι μονόγλωσοι. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν βοήθεια έτσι και έτσι γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα στον ξένο γιατρό και τον μονόγλωσσο ξένο βοηθό που γίνεται μέσω του συσκευή. Αυτό το έχουμε σε πολλές περιπτώσεις. Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι μας εντυπωσίασε το, αυτό που είπα και αυτό που είπατε. Έχω ταξιδέψει ολόκληρο τον κόσμο και με όλες αυτές τις ασκήσεις ένας από τους μεγαλύτερους μου φόβους είναι ακριβώς ότι ο κόσμος μπορεί να φοβάται να μιλήσει σε ένα μικρόφωνο ή σε μια τέτοια συσκευή. Από ό,τι φαίνεται όχι, δεν φοβούνται. Δεν έχουν ε, υγειονομική περίθαλψη, δεν έχουν εκπαίδευση, παιδεία. Όλοι έχουν όμως κινητά. <laughs> Το κινητό έχει τόσο πολύ δυσδύση στη ζωή την καθημερινή που το να μιλήσει κανείς σε ένα μηχάνημα δεν φαίνεται παράξενο στους λαούς του κόσμου. Ο κόσμος αλλάζει λοιπόν με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί οι φόβοι αυτής της φύσης, δηλαδή, να εξαλειφθούν σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ και η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σκοβρόσκι από το Πανεπιστήμιο του Πόζαν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Βάιβερ για την καταπληκτική του παρουσίαση και να εκφράσω την πεποίθηση ότι σίγουρα στο μέλλον τέτοιου είδους ε, εφαρμογέ θα χρησιμοποιούνται ευρέως. Αλλά να μην ξεχνούμε και ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα, μια κοινωνική πτυχή. Όταν έχουμε την εφαρμογή του συστήματος Bidula, του συστήματος αυτού. Πολύ συχνά, δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται σωστά αυτό το σύστημα μετάφρασης, ε, το σύστημα με τη βαλίτσα, το Bidula. Και μερικές φορές αντικαθιστά την ταυτόχρονη διερμηνία. Και, ε, και τέτοιες περιπτώσεις για τον ε, διερμηνέα της ταυτόχρονης μετάφρασης είναι σημαντικό και το θέμα της αποστολής. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η εφαρμογή τέτοιου συστήματος του βαλής είναι περιορισμένη και σε καμία περίπτωση ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέω όταν δεν εξασφαλίζει τεχνικέ προποθέσει και σίγουρα οι συσκευέ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο διερμηνέα. Um, yes, no I... Δεν μπορώ ε, συμφωνώ απόλυτα με το σχολείο σας και το κάνουμε διαρκώς αυτό. Γιατί όταν κάνουμε αυτές τις παρουσιάσεις θα διοικηθούμε σε απογοήτευση αν πιστεύουμε και αν νομίζουμε πως, ε, μάλλον δώσουμε την εντύπωση πως όλα τα τεχνικά προβλήματα έχουν λυθεί, ότι έχουμε φτάσει στην τέλεια κατανόηση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε στις ασκήσεις ε, που παρακολουθούμε. Συνήθως έχουμε διερμηνείς εκεί αλλά όχι τόσο πολύ. Σε κάποιες από τις εικόνες που είδατε λοιπόν σε αυτές τις ασκήσεις, συνήθως υπάρχουν 5 με 10 διερμηνείς. Και είναι συνήθως αρχάρι, δεν είναι, καθο... δεν είναι έμπειροι σαν ε, τους διερμηνείς που έχετε εδώ. Μπορεί να υπάρχουν θέματα με την ποιότητα της διερμηνίας, ωστόσο οι γιατροί τους ε, προτιμούν γιατί κατανοούν καλύτερα τον πολιτισμό, ε, τη γλώσσα κτλ. Δεν αρκούν όμως, άρα χρησιμοποιούμε και αυτές τις συσκευές. Ε, ας πούμε στις, στους σταθμούς όπου γίνεται ο διαχωρισμός, όπου απλώς στέλνουμε τον κόσμο στον κάθε γιατρό. Εκεί δεν ενοχλεί, απλώς είναι ένα εργαλείο ένα εργαλείο και είναι και ένα παράδειγμα αυτό αυτή τη συμβίωση για την οποία μίλησα. Ναι, χρησιμοποιούμε έναν διερμηνέα, έναν άνθρωπο, ενώ τα θέματα ρουτίνας μπορούν να γίνουν κάλλιστα από ένα μηχάνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ευχαριστήσουμε θερμά τον ε, Δ. Βάιβελ για την ε, συναρπαστική παρουσίαση που μας έκανε. Y necesitamos Χρειαζόμαστε 1,5 λεπτό για να θέσουμε σε λειτουργία τις νέες τεχνολογίες και να δώσουμε το λόγο στον επόμενό μας ομιλητή. Bien. Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον επόμενο, τον μας καλεσμένο, έναν ερευνητή, τον δόκτωρα Χερβέ Άντελμαν, που είναι ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης και θα μας βυθίσει στο συναρπαστικό κόσμο του ανθρώπινου εγκεφάλου και το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός διερμηνέα στη διαδικασία της ταυτόχρονης διερμηνίας. Και μάλιστα θα μας πει τι θα συμβεί και στα ενιδρία. Τι γίνεται στα ενηδρία, στον εγκέφαλο των, εγκεφα... Ε, στον εγκέφαλο των διερμηνέων αυτή τη στιγμή που εργάζονται και ελπίζω να μην τρομοκρατηθούν οι διερμηνείς από αυτά που θα δουν και θα ακούσουν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω ιδιαίτερη χαρά και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ στην σημαντική αυτή ομίγυρη και ελπίζω να είναι εξίσου σημαντική και η δική μου παρουσίαση. Θα σας παρουσιάσω το έργο που, και τις έρευνες που κάνουμε στην ε, Γενέβη για την νευροεπιστήμη της, ε, της διερμηνίας και την ανάλυση της διερμηνίας. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε μια βιολογική προσέγγιση. Δεν πρόκειται φυσικά να ε, καταπολεμήσουμε ή να εξαφανίσουμε τη μαγεία της διερμηνίας, αλλά να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του διερμηνία, πώς μπορεί να μάθει κανείς αυτή τη, ε, την διεργασία, το έργο του διερμηνέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό και να σας πω γιατί ε, προσπαθήσαμε να ε, μελετήσουμε και να ερευνήσουμε αυτό το θέμα. Η διερμηνία είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι ένα έργο που προϋποθέτει τεράστια συγκέντρωση, ε, μεγάλες γλωσσικές γνώσεις και μπορεί να γίνει μετά από μακροχρόνια εξάσκηση και κυρίως πρακτική. Για μας η διερμηνία είναι εξαιρετικό μοντέλο για να εξηγήσουμε και τις βάσεις του γλωσσικού και γνωστικού ελέγχου και στη διάρκεια της εξάσκησης παρακολουθήσαμε ασκούμενους διερμηνείς ε, και το θέμα της πλαστικότητας του εγκεφάλου, δηλαδή πώς προσαρμόζεται ο εγκέφαλος στις λειτουργίες και τις ανάγκες αυτού του έργου που έχει να επιτελέσει. Όπως είπα και προηγουμένως, η γνώση της διερμηνίας δεν προϋποθέτει μόνο γλωσσικές γνώσεις. Αυτό το ακούσαμε και χθες όταν μιλήσαμε για την κατάρτιση των καλών διερμηνέων. Η διερμηνία είναι ένα έργο που γίνεται με πολλή δυσκολία ε, και κυρίως ε, θέματα αντίληψης, γιατί ο διερμηνέας αυτή τη στιγμή ακούει ταυτόχρονα εμένα και ταυτόχρονα ακούει το μήνυμα που αναπαράγει ο ίδιος. Ε, γι' αυτό έχω κάνει αυτή τη διαφάνεια, για να καταλάβετε. Αυτό συμβαίνει αν προσπαθεί κανεί να παρακολουθήσει ταυτόχρονα δύο γλώσσες με μια μικρή χρονική διαφορά. Επιπλέον, πέραν τούτου υπάρχουν και οι γλωσσικέ απαιτήσει. Ο διερμηνέα φυσικά θα πρέπει να εφομοιώσει το περιεχόμενο της, ε, ε, του μηνύματο και να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και μάλιστα σχετικά πιστά. Ελπίζω αυτό να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μαγικό που γίνεται μια τέτοια διαργασία. Επιπλέον, κάτι τέτοιο προϋποθέτει έναν έλεγχο πολλών ικανοτήτων, ικανότητα προσοχής, ε, γνωστικές επίσης ικανότητες. Θα πρέπει κανείς να ακούει συνέχεια με ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρωμένος και φυσικά να τα μεταφέρει όλα αυτά και χωρί λάθη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει μεγάλη ευελιξία του εγκεφάλου. Επίση, ε, ο εγκέφαλο των ε, δίγλωσσων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας. Ο εγκέφαλος των δίγλωσσων παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τις εκτελεστικές λειτουργίες. Δηλαδή, οι δίγλωσσοι έχουν καλύτερο έλεγχο της προσοχής, πολύ πιο εύκολα ε, μεταβαίνουν από το ένα στο άλλο έργο που γίνεται ταυτόχρονα και επίσης έχουν καλύτερη δυνατότητα ε, αναστολής. Όταν δηλαδή ξεκινούν μια χειρονομία ή μια ε, δράση, πολύ πιο εύκολα μπορούν να τη σταματήσουν ή να την περιορίσουν. Επίσης ε, υπάρχουν ε, μελέτες που δείχνουν ότι η δίγλωση διερμηνείς έχουν ένα γνωστικό αποθεματικό που τους προστατεύει από την παράνοια. Τα συστήματα της, ναι, άνοια. της ναι. άνοιας εμφανίζονται πολύ λιγότερο σε, θέμα, σε δίγλωση από τις ε, μονόγλωσσους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτή η προστασία από την άνοια για τους δίγλωσσους. Βλέπουμε εδώ, στο, στη γραφική αυτή απεικόνηση, τις ε, δημοσίευσεις που έγινε για τις εκτελεστικές και γνωστικές ε, λειτουργίες στους πολύγλωσσους τα τελευταία 15 χρόνια. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των δημοσιεύσεων είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και πολύ επίκαιρο. Εγώ θα περάσω τώρα στις νευροεπιστήμες και θα σας κάνω μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των, της γέννησης των νευροεπιστημών. Οι αρχές της νευροεπιστήμης ανάγονται στο 19ο αιώνα. Τότε υπήρχαν φρενολόγοι που υιοθετούσαν τη γνώμη ότι ο εγκέφαλος απαρτίζεται από διάφορα όργανα που το καθένα επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Και τα όργανα αυτά αντικατοπτριζόταν στην μορφή, στο σχήμα του εγκεφάλου. Έτσι μπορούσε κανείς ε, ψηλαφώντας τον εγκέφαλο να καταλήξει ορισμένα συμπεράσματα. Γνωρίζουμε ότι αυτό πια δεν... Το κρανίο, συγγνώμη, να καταλήξει συμπεράσματα. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτό σήμερα δεν ευσταθεί. Επίσης ε, δημιουργούσαν κάποιους δεσμούς μεταξύ των, ε, των ε, βλαβών του εγκεφάλου και κάποια, κάποιες συμπεριφορές. Εδώ έχουμε ένα πολύ γνωστό εγκέφαλο και το πορτρέτο ενός πολύ γνωστού επιστήμονα, του Πιερ Πολ Μπροκά. Εδώ έχουμε τον εγκέφαλο, έχουμε το προφίλ, έχουμε το εμπρόστιο αριστερό τμήμα και το πίστιο δεξί, και ο Πιέρ Μπροκά είχε έναν ασθενή των Λεμπόν που ήταν ανίκανος να προφέρει οτιδήποτε άλλο από την συλλαβή Ταν. Ε, μετά το θάνατο του ασθενούς αυτού διαπιστώθηκε ότι είχε μια εγκεφαλική βλάβη στην περιοχή αυτή που έχει πάρει πια το όνομα του Μπροκά, ονομάζεται περιοχή Μπροκά. Βρίσκεται στον ε, μετωπιαίο λοβό και είναι μια περιοχή που ε, όταν κανείς ακούει τους ήχους, ε, κάνει την κατανομή των ήχων. Ο ασθενής αυτός μόνο ταν μπορεί να κάνει, γιατί δεν, μπορούσε, δεν είχε παραστάσεις από άλλα φωνήματα. Παρ' όλα αυτά μπορούσε να καταλαβαίνει ότι άκουγε. Ε, αργότερα ο Καρλ Βέρνη και άλλος καθηγητής διαπίστωσε ότι ε, ασθενείς του με κεφαλικές βλάβες είχαν πολλά προβλήματα στην ομιλία και έκανε εργασίες ε, κυρίως στην περιοχή που σήμερα έχει πάρει το όνομά του, την περιοχή Βέρνικε, μία περιοχή που ασχολείται με την αντίληψη, την κατανόηση της ομιλίας. Και οι ασθενείς του Βέρνικε δεν μπορούσαν να καταλάβουν μία ομιλία, αλλά ταυτό, ε, ενώ μπορούσαν να μιλήσουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και λάθη. Οπότε έχουμε μία αποσύνδεση μεταξύ της κατανόησης του λόγου και της εκφοράς του λόγου. Άρα τα τμήματα του εγκεφάλου που χειρίζονται τις δύο αυτές λειτουργίες είναι διαφορετικά. Λίγο αργότερα ακόμη είχαμε έναν γνωστό νευροχειρουργό, τον Βίλτερ Πένφιλτ, που ε, μελέτησε ζωντανού ανθρώπου, γιατί όταν έκανε χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο χρησιμοποιούσε ηλεκτρική διέγερση έβαζε ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο των ασθενών του. μάλιστα δεν υπάρχουν ε, αισθητήρε πόνου στον εγκέφαλο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει σε αναισθησία, ε, υπό αναισθησία αυτή η ασθενή. Και ε, ενδιαφέρθηκε κυρίως για τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τις αισθήσει και για τις κινητικές λειτουργίες. Και τότε περάσαμε από την ε, έρευνα και τις μελέτες ε, σε νεκρούς ε, ε, στην έρευνα σε ζωντανούς. Έχουμε φυσικά πολύ λιγότερο επεμβατικές πια τεχνικές και θα σας παρουσιάσω την πιο σύγχρονη. Εδώ έχουμε έναν μαγνητικό τομογράφο. Επικόνηση με μαγνητική τομογραφία που μας δίνει πολύ ωραίες και πιστές εικόνες του εγκεφάλου, όχι μόνο του διαρθρωτικού τμήματος αλλά και του λειτουργικού τμήματος. Και θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Εδώ θα δείτε δύο σύντομες ταινίε από ε, που έχουν περάσει από μαγνητικό τομογράφο. Βλέπετε εδώ το μέσο του εγκεφάλου και βλέπουμε τι γίνεται από την επιφάνεια μέχρι το κέντρο του εγκεφάλου, χάρη στην ε, τεχνική αυτή της μαγνητικής τομογραφίας. Και εδώ έχουμε έναν εγκέφαλο που περιστρέφεται γύρω από τον κάθετο άξονά του. Εδώ έχουμε την μορφολογία του εγκεφάλου, αλλά έχουμε και πολύ πιο εκλεπτισμένες εικόνες. Για παράδειγμα, τη συνδεσιμότητα. Εδώ βλέπουμε ε, μακαρονιών κάπως ε, ρευστή εικόνα. Εδώ έχουμε τις διάφορες περιοχές, ε, την καλωδίωση αν θέλετε του εγκεφάλου. Έχουμε μια περιοχή που είναι υπεύθυνη για την κατανόηση και άλλη που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του λόγου, της ομιλίας. Εδώ μπορούμε να, να εξετάσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου. Εδώ έχουμε δύο αισθητηριακέ λειτουργίες, αισθητικές λειτουργίες. Ε, στη μία περίπτωση έχουμε αντίδραση σε ένα απλό ε, ε οπτικό ερέθισμα και βλέπουμε ότι στον ινιακό λοβό, στον ε, ε, οπτικό εγκεφαλικό φλοιό έχουμε την αντίδραση. Και εδώ έχουμε ε, ακουστική διέγερση, ένας εγκέφαλος δηλαδή που ακούει φράσεις και βλέπουμε εδώ ότι ενεργοποιείται ε, ο κροταφικός λοβός και θα το δούμε αυτό καλύτερα στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος απορτίζεται από διάφορες περιοχές που επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να καταλήξουμε στην περίπλοκη συμπεριφορά που παρατηρούμε καθημερινά. Εδώ βέβαια είναι μια απλή απεικόνηση μιας εικόνας του εγκεφάλου και έχουμε τους διαφόρους λοβούς. Κάθε λοβός έχει διαφορετική λειτουργία. Έχουμε τον ενιακό λοβό που είναι υπεύθυνο για την όραση Έχουμε τον βρεγματικό, τον κίτρινο που χειρίζεται τις αισθητικές πληροφορίες. Έχουμε τον κροταφικό λοβό, σας τον ανέφερα πριν από λίγο, που είναι υπεύθυνο για την ακοή, τα συναισθήματα και τη μνήμη και έχουμε και το μετοπίο λοβό, που είναι η πιο ε, τελευταία, το πιο, το πιο σύγχρονο του μετοκεφάλου, το πιο πρόσφατο και ασχολείται με τις εκτελεστικές λειτουργίες, ε, τις γνωστικές λειτουργίες, την κίνηση, διαχείριση της σκέψης, το κόκκινο τμήμα. Ε, βέβαια, εμείς στις έρευνές μας ε, ενδιαφερόμαστε κυρίως για το μετοπιό και τον κροταφικό λοβό, γιατί αφορούν την, την ακοή, την διαχείριση των γνώσεων και την παραγωγή της ομιλίας. Τώρα, ποιες είναι οι νευρονικές βάσεις της ταυτόχρονης διερμηνίας και πόσο επηρεάζει η εμπειρία της διερμηνίας στη δομή και τις λειτουργίες του κεφάλου. Εμείς στη μελέτη μας παρακολουθήσαμε δύο ομάδες ασκουμένων διερμηνέων που παρακολουθούσαν το μάθημα διερμηνής στη Γενέβη και μία ομάδα ελέγχου με πολύγλωσσους φοιτητές σε σπουδές όμως που δεν είχαν σχέση με τις γλώσσες. Στην Γενέβη μάλιστα είναι τόσο κοσμοπολίτικο μέρος που έχουμε πολύ εύκολα βρίσκουμε πολύ εύκολα πολύγλωσσους φοιτητέ που δεν σπουδάζουν ιδιαίτερα γλώσσα, αλλά μπορούν εύκολα να μεταφράσουν απλές φράσεις. Οπότε προσπαθήσαμε να μελετήσουμε ε, τις συμπεριφορές των ασκουμένων ε, διερμηνέων και του, της ομάδας του ελέγχου στην αρχή στους 0 μήνες και μετά από 15 μήνες ε, τους ζητήσαμε να πραγματοποιήσουν τις ίδιες διεργασίες ε, μετά από 15 μήνες. Βέβαια δεν είναι ε, και πολύ ευχάριστο να μπει κανεί στον ε, μαγνητικό τομογράφο. Είναι σαν να μπαίνει σε μια σύραγγα και μάλιστα δημιουργείται και ένας τεράστιος θόρυβος, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε το έργο που ζητούμε από τους διερμηνείς και την ομάδα ελέγχου στις συνθήκες αυτές. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μεταφράσει συνεχόμενες, συνεχείς ομιλίες, αλλά με μονομένες φράσεις που αν τις συνθέσουμε δημιουργούν μια ομιλία, αλλά είναι κατακαιρματισμένες. Ακριβώς λόγω του θορύβου έπρεπε να κόψουμε τις φράσεις στην ομιλία. Αλλά δημιουργούμε ε, παρόλα αυτά ένα πλαίσιο της ομιλίας. Τώρα, προσπαθώντας να ε, αναλύσουμε τη λειτουργία της διερμηνίας, καταλήξαμε σε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Έχουμε την αντίληψη, την κατανόηση, την παραγωγή του λόγου, ένα είδος αυτοεπίβλεψης, δηλαδή ε, κανείς ελέγχει την παραγωγή του λόγου και επίσης ε, ταυτόχρονη διαχείριση δύο γλωσσών. Βέβαια, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες. Εμάς μας, μας ενδιαφέρει να ταξινομήσουμε τα χαρακτηριστικά της διερμηνίας, δηλαδή μηχανικές ε, χειρονομίες, αντίληψη, πράξη ε, αντίληψης ε, κατανόησης και αυτοελέγχου ή λιγότερο ενδιαφέρουσε από την ε, ταυτόχρονη διαχείριση δύο γλωσσών. Βέβαια, όλα είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτέλεση της διερμηνίας, αλλά προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το ρόλο των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου, συγκρίνοντας τη διερμηνία και ένα πιο απλό έργο, το σάντο, την διαδοχική επανάληψη φράσεων στην ίδια γλώσσα όμως, χωρίς διερμηνεία, δηλαδή. Επίσης κάναμε ένα βασικό έλεγχο ε, επιτρέποντας τους ε, φοιτητές μας να ακούσουν φράσεις και να δούμε πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλο σε, μια ακουστική διέγερση. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα στον εγκέφαλο που ενός ανθρώπου απλώ ακούει φράσεις. Βλέπετε ότι υπάρχει διμερής έντονη δραστηριότητα στον κροταφικό λοβό, κάτι που ανταποκρίνεται στις ε, ε, προσδοκίες μας, ότι δηλαδή ο εγκέφαλος ακούει και κάνει μια ανάλυση του λόγου. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον. Περνάμε σε μια, σε μια πιο απαιτητική εργασία που είναι η επανάληψη φράσεων. Εδώ βλέπω μια πολύ πιο έντονη κεφαλική δραστηριότητα. Και βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της ε, ταυτόχρονης ε, επανάληψης των φράσεων. Εδώ έχουμε όχι τις περιοχές που ασχολούνται με την ακοή, αλλά με τη διαχείριση του έργου αυτού. Βλέπουμε εδώ το τη δραστηριότητα από την επιφάνεια μέχρι το κέντρο και βλέπετε την έκταση αυτής της δραστηριότητας. Δεν καλύπτει μόνο την ε, επιφάνεια του εγκεφάλου, αλλά φτάνει μέχρι το κέντρο. Είναι δύσκολο επειδή κινούνται εικόνες να σας εξηγήσω. Προτιμώ μια στατική απεικόνηση. Εδώ στα δεξιά έχουμε εγκάρσιες τομές του εγκεφάλου και βλέπετε κάθετες ε, τομές και βλέπετε τις ε, περιοχές της κινητικής λειτουργίας που ασχολούνται με την παραγωγή του λόγου και με τη διαχείριση των χειρονομιών. Και αυτό φυσικά είναι σημαντικό για τη λειτουργία αυτή. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικές περιοχές. Στο μέσο του εγκεφάλου μια πολύ σημαντική περιοχή συνδέεται με τον έλεγχο της προσοχής και με την ανείχνευση των λαθών είναι μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιείται όταν διαπιστώνουμε ότι κάναμε ένα λάθος. Αυτή η περιοχή ε, ενεργοποιείται. Είναι σημαντικό να ακούει κανείς αυτό που λέει και να μπορεί να το ελέγχει και να διορθώνει το λάθος. Εδώ έχουμε μια οριζόντια τομή που δείχνει τους βαθύτερους πυρήνες στο κέντρο του εγκεφάλου, ε, στην περίπτωση της άρθρωσης η περιοχή αυτή που δημιουργεί ένα Β, ένα Β, μάλλον, είναι πολύ σημαντική περιοχή και είναι υπεύθυνη για τη βασική αντίληψη, τη στοιχειώδη αντίληψη και κυρίως τη διαχείριση των κινητικών λειτουργιών για να μπορεί κανείς να κάνει ε, πολύ πιο ε, ομαλές κινήσεις ε, και όχι απότομες και ξεκομμένες. Τώρα, τι γίνεται με την ταυτόχρονη διερμηνία έχουμε τον εγκέφαλο με τις ενεργοποιημένες περιοχές για τις, ε, την επανάληψη των φράσεων και με κόκκινο βλέπουμε τις περιοχές που ενεργοποιούνται με τη διερμηνία. Βλέπουμε ότι είναι ένα δίκτυο που εμφανίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά. Το αριστερό ημισφαίριο ενεργοποιείται κυρίως με την ε, διερμηνία και αυτό δεν μας εκπλήσει γιατί γνωρίζουμε ότι το αριστερό ημισφαίριο είναι αυτό που διαχειρίζεται τις πιο απαιτητικές λειτουργίες του λόγου, δηλαδή διαχείριση συντακτική και σημασιολογική. Δίνουμε τώρα τις ίδιες τομές, αλλά βλέπουμε σε κόκκινο χρώμα τις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται ιδιαίτερα με την ταυτόχρονη διερμηνία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε εδώ, σε αυτή την τομία αναριστερά την περιοχή Μπροκά. Αυτή ενεργοποιείται. Γιατί δεν διαχειρίζεται μόνο τη φωνολογία, αλλά καλύπτει και τη διαχείριση και την αντίληψη τα, της σημασιολογίας. Και εδώ κάτω έχουμε ένα τμήμα του μετοπιαίου λοβού που κάνει τη συντακτική επεξεργασία. Αυτό δείχνει ότι οι διερμηνείς που κάνουν αυτή την ε, λειτουργία προβαίνουν σε μια πολύ πιο βαθιά κωδικοποίηση των φράσεων. Πιο κάτω βλέπουμε ακόμη πιο ενεργοποιημένη δραστηριότητα στην περιοχή ε, αυτής της, ε, της, της ακοής, της, του ελέγχου και των, της, του εντοπισμού των λαθών και αριστερά βλέπουμε ότι στο κέντρο του εγκεφάλου είναι δύσκολο γιατί πρόκειται για ένα πολύ μικρό πυρήνα. Έχουμε τον κερκοφόρο πυρήνα που βρίσκεται στο επίκεντρο του εγκεφάλου και είναι μια περιοχή που διαχειρίζεται πολλές λειτουργίες. Για παράδειγμα, την κίνηση, τις κινητικές λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα την επιλογή, ε, την ε, επιλογή των κινήσεων και την ε, αναχέτηση μερικές φορές των κινήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το δίκτυο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γλωσσικό από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και εκτελεστικό. Έχει και πολύ γενικές λειτουργίες που επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της γνώσης. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο ποιες περιοχές του κεφάλου γενικά ενεργοποιούνται όταν κάνουμε αυτές τις λειτουργίες, αλλά ποιες είναι οι περιοχές του εγκεφάλου που διαχειρίζονται ε, αυτήν, ε, το input και το output τη στιγμή της διερμηνίας, δηλαδή την, ε, το άκουσμα της φράσης και την αναπαραγωγή στην άλλη γλώσσα. Και μάλιστα σε σχεδόν ταυτόχρονα. Ένα έργο που είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Έτσι λοιπόν καταμετρήσαμε τη διάρκεια της περίοδου ταυτοχρονισμού για κάθε φράση που ο κάθε φοιτητής έπρεπε να μεταφράσει και μετά εξετάσαμε το, το τμήμα του κεφάλου που επηρεάστηκε και που άλλαξε. Βλέπουμε ότι όσο, πιο όσο περισσότερο διαρκεί ο ταυτοχρονισμός, ο ταυτόχρονος χαρακτήρας της διερμηνίας, τόσο μεγαλύτερο τμήμα το κεφάλου επηρεάζεται. Βλέπουμε τι γίνεται εδώ στον ε, εγκεφαλικό φλοιό. Όταν έχουμε μια περίοδο ταυτοχρονισμού και κρατάει λίγο, έχουμε αυτή την εικόνα. Αλλά κάτι που συμβαίνει πιο κάτω είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε δύο μικρά τμήματα στο κέντρο που ενεργοποιούνται ανάλογα με τη διάρκεια αυτής της περίοδου του ταυτοχρονισμού. Αυτό είναι το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα και μαζί με τον κερκοφόρο πυρήνα που σας ανέφερα προηγουμένως επιτρέπουν την αναχέτηση των χειρονομιών ή των ε, δράσεων που κάνουμε. Δηλαδή, όταν χρειάζεται να διαχειριστούμε ταυτόχρονα πολλές γλώσσες, θα πρέπει να εμποδίσουμε μερικές φορές μία, ε, μία δράση για παράδειγμα, έχουμε πολύ διαφορετική λειτουργία από ότι όταν απλώς επαναλαμβάνουμε μία φράση. Τώρα προσπάθησα εδώ να κάνω μία διάκριση των περιοχών του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε αυτή τη διεργασία και εδώ δεν έχουμε πραγματικές δραστηριότητες. Έχουμε το δίκτυο ε, για την άρθρωση, την παραγωγή του λόγου, κυρίως ε, κινητικές περιοχές του εγκεφάλου Επίσης βλέπουμε εδώ ζώνες ε, για την ανείχνευση του λάθους, την επίβλεψη δηλαδή της ε, παραγωγής της ομιλίας και πλέον προσθέτουμε περιοχές που φαίνεται ότι εμπλέκονται στη διαχείριση του multitasking, της πολλαπλής ε, διαργασίας. Εκεί έχουμε ταυτόχρονη διαχείριση πολλών διαργασιών, πολλών εντολών. Αυτό γίνεται με ζώνες κυρίως ε, του μετοπιαίου λόγου. Και τώρα εδώ προσθέτουμε και την μετάφραση. Κάπως χονδρικά τα κάνουμε όλα αυτά. Έχουμε την περιοχή Μπροκά ε, και επίσης αυτή την περιοχή του κάτω μετοπιαίου λόγου και το κερκοφόρο πυρήνα στο κέντρο του εγκεφάλου. Τώρα, τι γίνεται σε ό,τι αφορά την επιλογή των διαφόρων ε, εναλλακτικών λέξεων όταν καλούμαστε να μεταφράσουμε μία γλώσσα. Εκεί ταυτόχρονα ενεργοποιούνται διάφορες περιοχές, γιατί χρειάζεται να μένουν ενεργές δύο γλώσσες. Εδώ περιστρέφουμε λίγο τον εγκέφαλο για να δούμε πώς είναι κατανεμημένες οι διάφορες περιοχές. Εδώ βλέπετε μια απεικόνιση τι συμβαίνει στο μυαλό του διερμηνέα που έχει εξασκηθεί στη διερμηνία. Σε φοιτητέ λοιπόν που έχουν αποφοιτήσει και τι γίνεται μετά από 15 μήνε όταν τελειώνουν τι σπουδέ του. Βέβαια δεν είναι επαγγελματίε ακόμη διερμηνεί γιατί χρειάζονται και πρακτική εξάσκηση. Αλλά έστω και μετά από 15 μήνε εξάσκηση ήδη διαπιστώνουμε αλλαγέ στον εγκέφαλο. Εδώ βλέπουμε τι λειτουργικέ αλλαγέ όταν ε, εξετάζουμε μετά από 15 μήνες, μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές, βλέπουμε τι συμβαίνει. Σε αυτές τις τρεις περιοχές του εγκεφάλου παρατηρούμε μία μείωση του επίπεδου της δραστηριότητας που απαιτείται για την παραγωγή του ίδιου έργου. Δηλαδή, ε, ο εγκέφαλο έχει γίνει πιο αποτελεσματικό, δεν χρειάζεται να κινητοποιείται τόσο πολύ, να ενεργοποιείται τόσο πολύ μετά του 15 μήνες. Και βλέπουμε εδώ δεξιά έχουμε πάλι τον κερκοφόρο πυρήνα και όπως σας είπα, ο πυρήνας αυτός ασχολείται με τη διαχείριση της γνώσης, ε, των κινητικών λειτουργιών και δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την ομιλία. Η μόνη περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην ομιλία είναι αυτή η περιοχή που συνδέεται με την κατανόηση και την ε, συντακτική διαχείριση, με την στοιχειώδη ουσιαστικά κωδικοποίηση του περιεχομένου των φράσεων. Πέραν των λειτουργικών λοιπόν αλλαγών, διαπιστώνουμε και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στον εγκέφαλο μετά από 15 μήνες εξάσκηση. αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ότι μέσα σε 15 μήνες ε, αλλάζει ο εγκέφαλος. Εδώ βλέπουμε το ε, τις δραστηριότητες σε γαλάζιο και κίτρινο χρώμα και βλέπουμε τις ζώνες που έχουν αλλάξει μετά την 15μηνη ε, αυτή εξάσκηση. Αλλάζει ο όγκος κάποιων δομών του εγκεφάλου. Και βλέπουμε πυρήνες ε, στο κέντρο του εγκεφάλου, που είναι αυτοί που εμπλέκονται περισσότερο, το κερκοφόρος πυρήνας, ε, έλυφος του φακοειδούς πυρήνα, και που εμπλέκονται στην διεργασία και αλλάζει ο όγκος τους. Και μάλιστα αυτές οι περιοχές είναι γνωστικές, γενικές γνωστικές περιοχές, δεν είναι καν γλωσσικές περιοχές. Οπότε η εξάσκηση αυτή στη διερμηνία έχει αλλάξει ριζικά τη μορφή ε, του εγκεφάλου και τη διάρθρωση και την λειτουργία. Και δεν ξέρω τι διαφορές θα έχει και στην καθημερινότητα πέραν της ε, των διαφορών στις γνωστικές λειτουργίες. Αυτά λοιπόν και σας παρουσιάζω εδώ τις συνεργάτηδές μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου, το πολύ δεκαπέντε λεπτά για έρωτα αποκρίσεις. Νομίζω η Κλέρ Ντόνοβαν θέλει το λόγο από τον ΩΣΑ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό και επίσης ε, ικανοποιητικό για να βλέπουμε οι διερμηνείς ότι έχουμε ε, μια ενίσχυση των γνωστικών περιοχών και μια προστασία κατά της άνοιας. Αν και δεν είμαι και βεβαία, εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το κεντρικό μου θέμα, πάντως ήθελα να ξέρω αν έχετε την πρόθεση να κάνετε μελέτες ε, σε έμπειρους διερμηνείς που έχουν πολλά χρόνια πείρας, γιατί συχνά έχω διαπιστώσει ότι μετά από 2-3 χρόνια Επαγγελματική πείρα, οι διερμηνείς ε, δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Ε, γίνονται πραγματικά έμπειροι ξεπερνούν τις αρχικές τους γνώσεις. Έπειτα θα ήθελα να ξέρω αν πιστεύετε πως μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες του θορύβου μέσα στα σκάνερ για να μπορείτε να δείτε συνεχείς ε, ομιλίες. Γιατί φαντάζομαι ότι θα ενισχυθούν όλα αυτά τα στοιχεία αν υπάρχει μια κανονική ομιλία και όχι μόνο απομονωμένε φράσεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που μπαίνουν σε λειτουργία σίγουρα, όπως η πρόβλεψη κτλ. Και έπειτα να δούμε αν υπάρχει κινητοποίηση των περιοχών που διαχειρίζονται τις συστήσεις, τα συστήματα, γιατί με ενδιαφέρει πολύ για την ε, παιδαγωγική. Σας ευχαριστώ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Ε, ναι, τώρα κοιτάμε, εξετάζουμε κυρίως τους πιο έμπειρους ε, διερμηνείς και θα θέλαμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα στους ίδιους διερμηνείς που παρακολουθήσαμε γιατί μία τέτοιου είδους μελέτη έχει συνήθως ενδιαφέρον. Σε σχέση με τα όσα λέτε για την μέθοδο εργασίας που αλλάζει στους έμπειρους διερμηνείς, Σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω και υποψιάζομαι ότι οι περιοχές οι οποίες μηχανικά εμπλέκονται στην διερμηνία δεν θα αλλάξουν πολύ, γιατί αυτό που διαπιστώνουμε είναι μία μείωση της δραστηριότητας αυτών των περιοχών. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή με την εμπειρία το εγκέφαλος γίνεται πιο αποτελεσματικός και διαχειρίζεται το έργο αυτό με μεγαλύτερη ευκολία. Αν δούμε κάτι δηλαδή μάλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Έχω την εντύπωση. Τώρα όσον αφορά τη δομή θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν η μείωση τη δραστηριότητα συνοδεύεται και από διαρθρωτικές αλλαγέ στο γνωστικό, στις περιοχές. Τώρα για το θόρυβο και τι δυσκολίε που έχουμε το σκάνερ έχουμε πρόβλημα. Ναι, το ένα είναι ο θόρυβο και το άλλο είναι ότι η μαγνητική τομογραφία είναι μια τεχνική που μα δίνει εικόνε. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν τεχνικέ που μα επιτρέπουν να κάνουμε ε, σε, ε, με χιλιοστά των δευτερολέπτων ε, τις εικόνες. δύο εικόνες που είδαμε είναι κανείς δύο δευτερόλεπτα. Όταν, δύο δευτερόλεπτα όταν κανείς μιλά είναι πολύ χρόνος γιατί κινούμαστε πολύ όταν μιλάμε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ λίγες τεχνικές νευροαπεικόνσεις που να μας διευκολύνουν όσον αφορά την κίνηση. Έχουμε μόνο την τεχνική NILS που μπορεί να ε, βοηθήσει. Όμως δυστυχώς αυτή η τεχνική δεν μπορεί παρά να δει την παρά μόνο την επιφάνεια του εγκεφάλου, δεν, του φλοιού, δεν μπορεί να μπει σε βάθος. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Φυσικά θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον να τα καταφέρναμε, γιατί όντως υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Η πρόβλεψη όντως είναι κάτι που δεν καταφέρνουμε να δούμε με αυτές τις τομές. Τώρα για τα αισθήματα. Εμείς προσπαθήσαμε οι φράσεις μας να είναι πολύ ουδέτερες, ε, οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε τις, ε, τα συναισθήματα και αυτό για να αποφύγουμε την ύπαρξη πολύ ειδικευμένου λεξιλογίου και για να μην αποσπαστεί η προσοχή των διερμηνέων από το περιεχόμενο. Και μένα με ενδιαφέρει αυτό το στοιχείο πολύ, γιατί έχω την εντύπωση ότι η αυτόματη διαχείριση των συναισθημάτων είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι, και όχι μόνο οι διερμηνείς, δεν είμαστε σε θέση να σταματήσουμε την επεξεργασία των συναισθημάτων ε, ε μέσω, τα όσα βλέπουμε, τα όσα ακούμε, ένα θόρυβος, ε, μια φωνή. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συναισθηματικές μας, τα συναισθηματικά μας αντανακλαστικά και θέλω να δω αν οι διερμηνείς το καταφέρνουν τελικά αυτό. Αυτό που εγώ έχω διαπιστώσει στην ε, διδασκαλία, γιατί έχω διδάξει εδώ και 25 χρόνια, είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συναισθήματα μέσω της διαχείρισής τους, δηλαδή μια μερική αναχέτηση, μια αποστασιοποίηση, αλλά πάντως χρήση των συναισθημάτων, πράγμα που επιτρέπει καλύτερη κατανόηση του μηνύματος. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νικόλαη Μπορόφσκι ε, τώρα από τον Όσα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Έχω και μια ερώτηση γιατί κάνω στα ρωσικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα ε, λοιπόν να πω το εξή. Θα μπορούσα να ψάξω το διαδίκτυο για να ενημερωθώ, αλλά θα ήθελα να αξιοποιήσω τη δική σας παρουσία για να σας ρωτήσω το εξή. Υπάρχει καμιά ουσιαστική διαφορά ε, με βάση τις τελευταίες γνώσεις για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Υπάρχει καμιά θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε ε, διάφορες γλώσσες, μητρικές γλώσσες, ενώ όταν μαθαίνει κανείς όταν είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις ξένες λεγόμενες γλώσσες, αυτές που μαθαίνουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και σε ό,τι αφορά έτσι, τοπογραφικά τις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα ή μια γλώσσα την οποία έχει μάθει ε, το άτομο αργότερα και ε, κατά τη διάρκεια της διερμηνίας. Το έχετε μελετήσει αυτό και ποιες είναι οι συνέπειες. Δηλαδή και την προστασία από τη γεροντική άνοια, την ε, και τη λοιπά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίσω από την τελευταία για την άνοια. Δυστυχώς ε, δεν ε, έχει αποδειχτεί αυτό από τις δικές μου εργασίες, αλλά φαίνεται ότι η δίγλωση, το έχουν ε, αποδείξει αυτό στον Καναδά οι έρευνες, η δίγλωση ανεξάρτητα από τη γλώσσα είναι πιο προστατευμένη. Όταν χρησιμοποιεί κανείς δύο γλώσσες με τρόπο ενεργητικό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Υπάρχει εδώ ένα απόθεμα γνωστικό. Δηλαδή, ε, το, ο εγκέφαλος μπορεί να καταστραφεί από την όσο του Αλτσχάιμερ ή από άλλα νοσήματα αρκετά μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ε, άνοιας. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες. Ε, τώρα για το πώς αντιπροσωπεύονται οι γλώσσες ή πώς φαίνονται στον εγκέφαλο. Αυτό έχει προβληματίσει και συναρπάζει τους ερευνητέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μένα προσωπικά, αλλά δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση έτσι απλή και σύντομη. Όταν έχουμε δύο γλώσσες και χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο στους δίγλωσσους, ε, ε, ένας δίγλωσσος ισόρροπος, ας πούμε, στη χρήση του και των δύο γλωσσών, ε, δεν έχει διαφορά ε, στη χρήση της γλώσσας. Αντίθετα, όταν είμαστε σε διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας, υπάρχουν κάποιες περιοχές του εγκεφάλου που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση, υπησέρχονται και χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση και την επεξεργασία της γλώσσας. Και όσο προχωράει η πραγματογνωμοσύνη και η εμπειρία, τόσο ε, συμπλησιάζει η εικόνα. Δηλαδή, όταν κάποιος μαθαίνει μια δεύτερη, μια τρίτη γλώσσα, ο εγκέφαλος ε, λειτουργεί ε, με το δεξί ημισφαίριο. Προηγουμένως σας είπα πάρα πολύ σύντομα ότι είναι πιο έντονη η δραστηριότητα για τις γλώσσες στο αριστερό ημισφαίριο. Ενώ εδώ ε, πολύ διαφορετικές περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου χρησιμοποιούνται γνωστικές περιοχές για την εκμάθηση της γλώσσας, για τη σκέψη είναι μια ενεργή ε, γνωστική διαδικασία. Ενώ στη μητρική μας γλώσσα ή τη γλώσσα που κατέχουμε απόλυτα δεν υπάρχει ε, γνωστική ε, λειτουργία. Όλα είναι αυτόματα πάνω κάτω. Εκεί λοιπόν αρχίζει και επέρχεται μια αλλαγή, όταν γίνεται αυτόματη αυτή η χρήση. Ξέρω ότι η απάντησή μου δεν είναι ικανοποιητική, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα για τις ε, δομικές διαφορές του εγκεφάλου μεταξύ ε, ανθρώπων που χρησιμοποιούν μία ή δύο γλώσσες, γιατί είναι τόσο ετερογενής ο κέφαλος από άτομο σε άτομο, που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με τρόπο απόλυτο και με κατάλογο ε, των περιοχών. Γιατί ο λόγος είναι μια κίνηση, μια χειρονομία, αλλά χρειάζεται και ένα σημασιολογικό πεδίο κάθε φορά. Ε, χρειάζεται έννοιες, γιατί ε, κινητοποιούμε ας πούμε κάποιους τομείς για το χέρι, για να κουνήσουμε το χέρι μας. Αυτό ε, προέρχεται από διάφορες περιοχές του κεφάλου, είναι πάρα πολύ διάχυτη εικόνα. Αν είχαμε μία γλώσσα που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο είδος λεξιλογίου, θα μπορούσαμε να το μελετήσουμε. Αλλά αυτά είναι υπερφυσικά, δεν είναι φυσιολογικά, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν. Ευχαριστώ. Τρεις ακόμα θέλουν να κάνω ερώτηση και προτείνω μετά από τους τρεις αυτούς να κλείσουμε τον κατάλογο και να κάνουμε το διάλειμμα για το καφέ. Τον Φοκ από τον Άτομο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ συναρπαστική, ενδιαφέρουσα αυτή η ε, παρουσίαση. Έχω μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη απάντηση, απλώς παρατήρηση. ποιο ε, είναι το τμήμα του συνειδητού και του υποσυνείδητου σε έναν έμπειρο διερμηνέα. Ε, το έχετε μελετήσει τι γίνεται με τη γνώση και την πείρα. Επίσης έχετε μελετήσει ε, την απώλεια ορισμένων ικανοτήτων στους έμπειρους διερμηνείς. Είπατε τι κερδίζουν, χάνουν τίποτα. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Μόλις διάβασα το γυναικείο εγκέφαλο, the female brain. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι μάλλον φεμινιστής, αυτό ίσως θα μπορούσε να εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Και μία πρόταση για να αναπαραγάγουμε σε ένα τομογράφο το τι γίνεται στη διερμηνία. Μήπως να ζητήσουμε από τους υποψηφίους να μην εκφέρουν το λόγο, απλώς να φαντάζονται στο μυαλό τους τι θα έλεγαν. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, εξαιρετικές. Να αρχίσω με τη σειρά. Για το συνειδητό και το ασυνείδητο, δυστυχώς δεν έχω καμία απάντηση να σας δώσω. Οι εργασίες μας δεν μπορούν αυτό να το ε, διακρίνουν. Ε, ούτε έχω απάντηση για το αν μιλάνε, απλώς φαντάζονται οι διερμηνείς στη διερμηνία στον τομογράφο. Τώρα, ως προς την απώλεια ορισμένων ικανοτήτων. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φυσικά αλλά ε, ούτε εδώ είμαι σε θέση να σας δώσω σαφή απάντηση για τους διερμηνείς. Γνωρίζουμε ε, ότι ο εγκέφαλος ενός δίγλωσσου έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα. Για να βρει την κατάλληλη λέξη κάθε φορά, ο πολύγλωσσος έχει δυσκολία. Αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε και αποδεικνύεται. Ε, για να πει αν μια λέξη που βλέπει σε μια οθόνη υπάρχει πραγματικά ή δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν εξηγείται μόνο από τη διγλωσία ή την πολυγλωσία, είναι ότι έχει πολλέ γλώσσε στον εγκεφαλό σου και επιβραδύνεται αυτή η λειτουργία. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση μειονεκτήματο που έχω υπόψη μου. Βέβαια εξαρτάται και ε, από το περιβάλλον που κινείται κανείς όταν θα πρέπει να εκφράζεται με μεγαλύτερη ευχαίρεια μπορεί να είναι αυτό μειονέκτημα. Αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Για τους διερμηνείς θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Τώρα, από την άλλη, άκουσα ότι ορισμένοι διερμηνείς έχουν την εντύπωση ότι η μνήμη τους φθήνει ε, με την πάροδο των ετών. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Απλώς οι περιοχές του εγκεφάλου που ενέχονται κατά τη διάρκεια της διερμηνίας ε, μπαίνουν σε ένα δίκτυο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη φωνολογική ε, μνήμη. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα φανταζόμαστε τη φωνή που ακούμε είναι κείμενο που διαβάζουμε. Και εργαζόμενοι έντονα με αυτό το σύστημα δεν κινδυνεύει να φθήνει, απλώς εξειδικεύεται για μια πρακτική, για μια πολύ βαθιά μορφή κωδικοποίησης του περιεχομένου του μηνύματος. Ε, εκεί μπορεί να υπάρχουν λεπτές διαφορές, αλλά τώρα Ε, ας πούμε μπορεί να αποκλείεται η περίπτωση της αναγνώρισης ποιου μίλησε αυτά τα επιφανειακά. Τώρα το θέμα άνδρας γυναίκα είναι πάρα πολύ επίμαχο και δεν τολμώ σχεδόν να ε, αποφανθώ. Πρέπει να σας πω ότι οι ομάδες που μελέτησα ήταν ε, αρκετά ισορροπημένες από πλευράς φίλου άνδρες γυναίκες. Δεν έχω καμιά ειδική παρατήρηση. Και το τελευταίο για το θόρυβο στον τομογράφο. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και κάτι ακόμα. Η διερμηνία είναι μια χειρονομία. Είναι κάτι... Έπρεπε πραγματικά να γίνει διερμηνία. Δηλαδή έπρεπε κυρίως οι ε, συμμετέχοντες να ακούν τη φωνή τους. Γιατί αν δεν το έκαναν αυτό δεν θα μπορούσαμε να μελετήσουμε πρώτον εάν σωστά ε, διερμήνευαν. Εντάξει, τους εμπιστευόμαστε. Αλλά κυρίως για να δούμε τι γίνεται στον ε, εγκέφαλο και τι σημαίνει να είσαι υποχρεωμένος να ακούς τη φωνή σου. Γιατί εγώ είμαι δίγλωσσος και μπορώ να μεταφράσω, να διερμηνεύω ε, νοερά, αλλά στην πραγματικότητα για να μιλήσω δεν μπορώ να κάνω διερμηνία. Δηλαδή να ακούω ε, μια ομιλία και να ακούω και τον εαυτό μου την ώρα που τη μεταφράζω. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα τους υπόλοιπους δύο που θα δώσω τώρα το λόγο στην Όλγα Γόροβα από το Πανεπιστήμιο του Αστραχάν και ε, στην ε, κυρία από το Πανεπιστήμιο του Γκόλγοη να ε, κάνετε μία ερώτηση παρακαλώ, Κάστη, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη, διότι θα ήθελα πραγματικά στις 11 και 4 το αργότερο να κάνουμε διάλειμμα. Και θα παρακαλούσα και το προσκεκλημένο μας να απαντήσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Παρακαλώ, Όλγα. Σας ευχαριστώ θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που έχω να θέσω την ερώτησή μου στη γλώσσα μου. Και η, γλώσσα μου είναι, η ερώτησή μου είναι σύντομη. Όπως ξέρετε, ένας διερμηνέας κάνει μια δουλειά που είναι πολύ αγχωτική και επιπλέον ε, βάζετε τον άνθρωπο μέσα σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Δηλαδή, μέσα στο τομογράφο. Εγώ που πάσχω από κλειστοφοβία, άμα με βάλετε εκεί μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω, να διερμηνεύσω, μάλλον θα χάσω και τον κόσμο μου, δεν ξέρω που βρίσκομαι πιστεύετε πραγματικά αυτές οι συνθήκες ε, ε, επηρεάσαν τα αποτελέσματα των μελετών σας ή πιστεύετε ότι δεν έχει σημασία που βρίσκεται ο διερμηνέας στο μυαλό του, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο πάντα. Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας θα πρέπει να πω, ναι, όντως το περιβάλλον ενός τομογράφου είναι λιγότερο αγχωτικό από ότι η ίδια η καμπίνα, αλλά είναι αρκετά αγχωτικό γιατί είναι ένα ιατρικό περιβάλλον, είμαστε άνετα, αλλά εν πάση περιπτώσει μας περικυκλώνει ένας τεράστιος μαγνήτης, 300, ε, 300 φορές πιο δυνατός από το μαγνητικό πεδίο της ε, γης. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δουλεύουμε με το ίδιο σύστημα, τον κερκοφόρο πυρήνα και τα συστήματα, ε, τα περιοχέ τις περιοχές μάλλον που επηρεάζουν την κινητοποίηση, που επηρεάζονται από το στρες και το άγχος. Ε, αυτό είναι ε, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω πως ναι, όντως μπορεί αυτό να επηρεάσει αρνητικά το άγχος, ε, την ποιότητα της διερμηνίας και κυρίως στο επίπεδο της ε, ταυτόχρονης διαχείρισης των γλωσσών που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και σας ευχαριστώ και πάλι για την ερώτησή σας. Εγώ έρχομαι από την ε, από τον Galway. Είναι περισσότερο παρατήρηση αυτό που θα κάνω παρά ερώτηση. Ε, η έρευνά σας είναι πραγματικά συναρπαστική. Ελπίζω ότι στην τρίτη σύνοδο των Βρετάνων θα μπορώ να σας πω πού έχει βελτιωθεί η γνωστική ικανότητα. Γιατί εγώ αυτό μελετώ. Αν η κατάρτιση των διερμηνέων βελτιώνει και άλλες γνωστικές ικανότητες ε, για γνώσεις δηλαδή άλλου είδους. Έχουμε πολύ καλό ακροτήριο σήμερα εδώ. Εγώ έχω την ε, αίσθηση και την ε, πίστη ότι αν τον εκπαιδεύεις έναν, έναν διερμηνέα δεν του δίνει μόνο τα εργαλεία για να είναι διερμηνέα, αλλά του δίνει δεξιότητε για την επιβίωση, για τη ζωή του ολόκληρη. Πιστεύω πω οι δέκα φοιτητέ που παρακολουθούν αυτό τα μαθήματα θα βελτιωθούν και σε άλλου τομεί όπου δεν θα είχαν ασχοληθεί αν δεν είχαν κάνει τέτοιου είδου κατάρτιση. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχόλιο σα, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ βέβαια βεβαίως δεν ανήκω στον τομέα της κατάρτισης διερμηνέων, αλλά είναι πολύ καλό ε, το ότι αποτελεί αυτό, η διερμηνία τη βάση για γενικότερες αλλαγές αυτό που λέτε είναι σωστό και θα αναμένω τα αποτελέσματα της δικής σας έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αποχαιρετούμε τον δόκτωρα Ερβέ Άντερμαν και τον ευχαριστούμε για την παρουσίασή του και την παρουσία του. Προτείνω να είναι λίγο πιο σύντομο το διάλειμμα που είχαμε προβλέψει για το καφέ. 20 λεπτά και παρά 25 παρακαλώ ξεκινάμε. Ευχαριστώ πολύ.